el señor presidente. Buenos días, queridas amigas. Καλημέρα σας ε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι. Άρχεται η συνεδρίαση με το πρώτο μας σημείο σήμερα το πρωί, την έκθεση του κυρίου Deutsch για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ετήσια της έκθεση για το 2008. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή, τον Ταμάς Deutsch, για τέσσερα λεπτά. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.